Good Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρία Μακάβαν, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Περιβάλλοντος, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Είμαι πολύ ευτυχής ε, που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αργανώνεται αυτή η συνεδρίαση σε σχέση με τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ε, γιατί μέσω αυτών θα μπορέσουμε να υπεραμεινθούμε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απανταχού της γης περιλαμβάνονται στις βασικές ε, αρχές ε, ε, η ισότητα των φύλων, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής. Είναι τροφή για σκέψη λοιπόν και για σας που ασχολείστε τόσο με, τις, με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και προέρχεστε από τόσες χώρες και τόσες διαφορετικές υπήρου σήμερα εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε ε, και προσπαθούμε γενικώ να βρούμε την πολιτική συνένεση για την ανάπτυξη. Αυτό στέλνει ισχυρό μήνυμα προς τα έξω γιατί δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να προχωρήσει στο θεματολόγιο του 2030 για την βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, μαζί με την ε, κυρία Μακάβαν και όλη την υπόλοιπη ομάδα χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ και σας ευχαριστούμε για τη δουλειά δουλειά σας. Πώς είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε την ανάπτυξη μέσω ε, των διαφόρων στοιχείων. Ε, άνθρωποι, πλανήτης, εταιρικές σχέσεις ε, και ευημερία. Αυτά είναι οι λέξεις κλειδιά η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει δεσμευμένη ε, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ε, ένα σεβασμό των ε, συμφωνιών, κυρίως δε της, της συνθήκης των Παρισίων μαζί ή χωρίς τις ΗΠΑ. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι pacta sunt servanda, ότι θα πρέπει δηλαδή οι συνθήκες και να υλοποιούνται θα πρέπει, και αυτό κάνουμε, να βάλουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο της ε, δράσης μας, ε, τους πολίτες μας δηλαδή. Όσον αφορά την ευημερία, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να εμπλακούμε περισσότερο ε, και να εμπλέξουμε περισσότερο και την κοινωνία των πολιτών ε, στις διαδικασίες αυτές, γιατί μέσω της εμπλοκής της κοινωνίας των πολιτών θα μπορέσουμε και να φέρουμε νέες επενδύσεις και να ανοίξουμε νέους ορίζοντες. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας ότι κύριο στοιχείο είναι η αποφυγή ε, συγκρούσεων ε, και ταυτόχρονα βεβαίως πόλεμος σε δύο μέτωπα, στο μέτωπο της εκπαίδευσης και στο μέτωπο της, ε, της απασχόλησης. Θα πρέπει οπωσδήποτε να καταπολεμήσουμε και την, τις συγκρούσεις παντού και οπωσδήποτε την τρομοκρατία. Αυτό γίνεται μονάχα μέσα από την οικονομική και εκπαιδευτική ανάπτυξη. Χαιρετίζω λοιπόν την παρουσία σας, ε, την παρουσία σας εδώ, ε, εσάς ε, που θέλετε την υλοποίηση του θεματολόγιου του 2030 και που μάχεστε γι' αυτό. Και να ξέρετε ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πλήρως σας υποστηρίζει σε αυτές τις προσπάθειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα δώσω άμεσα το λόγο στην Πρωθυπουργό της Νορβηγίας, κυρία Έρνα Σόλμπεργκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Κύριε Ταγιάννη, σας ευχαριστούμε που οργανώσατε αυτήν την συνάντηση για ε, την βιώσιμη ανάπτυξη. Η συμβολή σας θα είναι κρίσιμη στην επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Πρέπει όλοι ως πολιτικοί ηγέτες να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Οι ευρωβουλευτές είναι σε θέση να επηρεάσουν και την εθνική πολιτική στις χώρες τους και τις πολιτικές δράσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό είσαστε ιδιαίτερα σημαντικοί. Κύριε Πρόεδρε, μετά, την, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η παγκόσμια αρχιτεκτονική ε, για την ειρήνη με επίκεντρο τα Ηνωμένα Έθνη άρχισε να διαμορφώνεται. Και όπως είπε ο Ντάκ Χάμερσουλτ, δημιουργήθηκαν ε, για να ε, σώσει τον, ε, την ανθρωπότητα από την κόλαση. Το 1951 ξεκίνησε ο πυρήνας ε, που οδήγησε στην σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ανθρακά ε, και Χάλιβα, η ΕΚΑΧ. Και σκοπός ήταν ο πόλεμος να καταστεί αδύνατος και έκτοτε η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει εξυπηρετήσει καλά την Ήπειρό μα. Έχει ενισχύσει την ειρήνη, τη δημοκρατία ε, στην Ευρώπη. Θέλουμε λοιπόν να σώσουμε από την κόλαση την ανθρωπότητα. Αυτό όμω είναι ένα έργο που ποτέ δεν τελειώνει. Θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε κάθε μέρα τη δημοκρατία και την ειρήνη και στην Ευρώπη και αλλού. Η συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και με περιφερειακές οργανώσεις ε, είναι πιο σημαντική τώρα από ποτέ. Στον διασυνδεδεμένο και παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας αντιμετωπίζουμε τις ίδιε προκλήσεις όπου και αν ζούμε. Την αλλαγή του κλίματο, τη μετανάστευση, ε, τον ε, βίαιο Όλα αυτά αποτελούν απειλή για όλους μας. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε ένα πολιτικό πρόγραμμα που μπορεί να καθοδηγεί τις προσπάθειές μας. Έχουμε τους βιώσιμους στόχους της χιλιετίας ε, που ε, ενέκριναν τον Σεπτέμβριο του 2015 οι ηγέτες 193 χωρών και έτσι μπορούμε να πετύχουμε η οικονομική, ε, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Οι στόχοι αυτοί δεν είναι κυρίως θεματολόγιο Ανθρωπιστική βοήθεια, Όλες οι χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένε της δική μου χώρας, έχουν ε, να κάνουν δουλειά σε εθνικό επίπεδο για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Ωστόσο, απαιτείται ανθρωπιστική βοήθεια στις πιο φτωχές περιοχές του κόσμου, καθώς και στις περιοχές με τις συγκρούσεις. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στις περιοχές που επηρεάζονται από κρίσεις και συγκρούσεις. Δεν επιτρέπεται να αφήσουμε τα παιδιά και τους νέους να μην ε, λαμβάνουν εκπαίδευση ή να μην έχουν ελπίδα. Η μετανάστευση είναι κάτι που αποτελεί σημαντική πρόκληση για την Ευρώπη. Θα πρέπει να ελέγξουμε τα σύνορά μας με σεβασμό ε, για τις θεμελιώδεις αρχές, ε, χωρίς να ξεχνάμε τις διεθνείς υποχρεώσεις μας. Γιατί τόσοι άνθρωποι επιλέγουν να κάνουν αυτό το επικίνδυνο ταξίδι προς την Ήπειρό μας και γιατί δεν παραμένουν εκεί που γεννήθηκαν. Όλοι γνωρίζουμε ότι μέρος ε, των αιτιών αυτών είναι ότι δεν υπάρχουν ε, θέσεις απασχόλησης και δεν υπάρχει ελπίδα στις περιοχές από τις οποίες προέρχονται. Κύριε Πρόεδρε, χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία, περισσότερη ολοκλήρωση, περισσότερη διασυνοριακή συνεργασία και περισσότερο εμπόριο, όχι λιγότερο. Ο οικονομικός προτεξιονισμός ε, είναι μια προσπάθεια να γυρίσει κανείς πίσω το ρολόι. Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η βιώσιμη στόχη της χιλιετίας είναι ο δικός χάρτης προς το μέλλον που θέλουμε. Προς έναν κόσμο χωρίς φτώχεια, χωρίς κλιματική αλλαγή. Κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι αυτό είναι ουτοπικό. Είναι δυνατόν όμως να το πετύχουμε εάν όλοι επιδείξουμε πολιτική βούληση και χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Θα πρέπει λοιπόν τα λόγια να τα κάνουμε πράξεις και 193 χώρες έχουν προσυπογράψει αυτούς τους στόχους. Αυτό σημαίνει ότι 193 χώρες πρέπει να εργαστούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Οι βουλευτές τους και οι και η πολιτική τους. Και να παραθέσω τα λόγια του Βάστα Χάβελ. Δεν αρκεί το όραμα, θα πρέπει να γίνει πράξη. Δεν αρκεί να κοιτάμε τα σκαλιά, θα πρέπει να ανέβουμε τη σκάλα. Θέλω λοιπόν να σας καλέσω να καλέσετε εσείς τις κυβερνήσεις σας και άλλους παράγοντες να καταβάλουν προσπάθειες και στο Ευρωκοινοβούλιο και στις πατρίδες σας και για θέματα που αφορούν την Ευρώπη αλλά και για τα θέματα που αφορούν όλον τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Mrs. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, ομιλία σας και είναι μεγάλη χαρά που συνεργαζόμαστε μαζί σα για το θέμα αυτό και είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη η σημερινή ημέρα. Έχουμε πάρα πολλέ συναντήσει ε, και συνεδριάσει και πραγματικά ε, προσβλέπουμε στη συνεργασία την περαιτέρω τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη χώρα σα την Νορβηγία. σα. ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική αυτή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα θα δώσω την Προεδρία, ε, τα ενία τη Προεδρίας σε καλά χέρια. Η πρόεδρο τη συζήτηση, θα είναι και η πρόεδρο τη Επιτροπή, η κυρία Λίντα Μακέβαν. Σα αφήνω λοιπόν και σας παραδίδω την Προεδρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας υπενθυμίσατε τη σημασία των βιώσιμων στόχων της χιλιετίας και την ε, σημασία της στήριξης των δεσμεύσεων από πλευρά της Ευρώπης των ε, περιβαλλοντικών στόχων παρά την αλλαγή στην αμερικανική πολιτική. Συνάδελφοι, πρωτού ξεκινήσουμε τη συζήτηση με το πάνελ, γιατί δυστυχώ είναι φρικτή η κίνηση στις Βρυξέλλες και έχουν καθυστερήσει και οι κύριοι ομιλητέ. Έχουμε ένα βίντεο όμως να προβάλλουμε ένα βίντεο το οποίο εξηγεί των στόχων, τους βιώσιμους στόχους, αναπτυξιακούς στόχους και γιατί βρισκόμαστε εδώ σήμερα. We can be. We must be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 Συνάδελφοι, είδατε το μήνυμα που προβάλλατε για τους στόχους της χιλιετίας, τους βιώσιμους στόχους ε, ανάπτυξης. Θα σας ελέγξω στο τέλος, να δω ποιος δεν πρόσφυγε. Για τους κύριους ε, μιλητέ. μου είπαν πει ότι θα καταφτάσουν το αργότερο πέντε λεπτά μετά την ομιλία τη Πρωθυπουργού. Αλλά έχουμε θέματα με την κίνηση σήμερα. Αν μου επιτρέπετε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Γι' αυτό λοιπόν ε, ήρθε πρώτα η Πρωθυπουργό. Γιατί είχα συνοδεία αστυνομικών και από ό,τι φαίνεται η αστυνομία καταφέρει να φτάνει πιο γρήγορα. So, the Prime Minister very kindly agreed that... Συμφωνεί ευγενικά η Πρωθυπουργό ε, να δεχτεί ερωτήσει, μια και ε, έχουμε λίγο χρόνο. Να σα θέσω εγώ την πρώτη ερώτηση. Πώ προετοιμάστε η χώρα σα για την υλοποίηση των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων, Γιατί πρέπει να ομολογήσω ότι όταν μιλώ στου συναδέλφου στην εθνική κυβέρνηση, ο κόσμο ήξερε τι ήταν οι στόχοι τη χιλιετία. Ήταν κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι για να του ε, πετύχουν οι χώρε. Αλλά σαν να μην ίσχυαν και για μας. Αλλά οι νέοι αυτοί οι αναπτυξιακοί στόχοι θα ισχύσουν και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παρακολουθήσουμε το, μέχρι τον Ιούλιο πώς έχει επιτευχθεί η υλοποίηση αυτών των στόχων. Τι κάνει λοιπόν η Νορβηγία, έχετε κάτι να μας αναφέρετε. Πέρσι Αναφέραμε στην πρώτη συνοδό του ΟΗΕ τι κάναμε λοιπόν στην Νορβηγία. Έχουμε διαιρέσει τους στόχους σε δύο κατηγορίες. Οι παγκοσμιοποιημένοι διεθνείς στόχοι, στους οποίους συμμετέχουμε με άλλες χώρες και αυτό αποτελεί τμήμα της, εξ... Ε, πολιτικής, της εξωτερικής μας πολιτικής και της αναπτυξιακής μας πολιτικής και κάποιες μας από αυτούς τους στόχους μα ενδιαφέρουν ο ιδιαίτερω. Για παράδειγμα, για την δασοκομεία, για την αλλαγή του κλίματο, έχουμε αυτό το πρόγραμμα όπου πληρώνουμε για τα τροπικά δάση προσπαθούμε να συμμετάσχουν όσο πιο πολλές χώρες και αυξάνουμε όσο μπορούμε τις ε, δυνατότητές μας γιατί οι ωκεανοί στη χώρα μας καλύπτουν πολύ μεγάλη έκταση. Γι' αυτό λοιπόν ε, η διατήρηση των ωκεανών καθαρών είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος και παρακολουθούμε φυσικά τα αναπτυξιακά προγράμματα. Και κυρίως μας ενδιαφέρει το θέμα της εκπαίδευσης των κοριτσιών, της γενικότερης ισότητας. Μας απασχολούν πολύ τα θέματα αυτά. αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε όλα μας τα Υπουργεία, έχουμε εξετάσει τους 17 στόχους και έχουμε αποφασίσει ποιο Υπουργείο είναι αρμόδιο γιατί γίνονται σχετικές ε, εκθέσεις. Έχουμε 17 στόχους, αλλά 100 και πλέον ε, συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένε υποκατηγορίε. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιο είναι αρμόδιο γιατί. Για παράδειγμα, στην υγεία. Ναι, τα πάμε καλά σε ό,τι αφορά τι γεννήσει. Ε, είναι πολύ καλή η μητρική και η βρεφική υγεία, αλλά η ψυχική υγεία δεν είναι καλή στην Νορβηγία. Εντάξει, μετά από κάποια με σκι τα πηγαίναμε καλά και είμαστε πρώτοι. Είμαστε πρώτοι στην ευτυχία, γενικότερη, το γενικότερο επίπεδο ευτυχία στη ζωή, αλλά 500 από τα άτομα κάθε χρόνο από τους, τα 5 εκατομμύρια ε, αυτοκτονούν. 75% για παράδειγμα των ε, μαθητών συνεχίζουν την φίτηση στα σχολεία, αλλά 25% έχουν προβλήματα, ψυχικά προβλήματα συχνά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τα θέματα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι οι βιώσιμοι αναπτυξιακοί στόχοι κάνουν όλες τις χώρες να συμπεριφέρονται σαν αναπτυσσόμενε χώρε. Γιατί όλοι έχουμε τομεί στου οποίου δεν έχουμε πετύχει του στόχου μα και θα πρέπει να του πετύχουμε. Αυτό έχει γίνει συστηματικά μέσω των διαφόρων υπουργείων. Και προσπαθούμε να δούμε σε ποιου τομεί θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μα. Για να μπορούμε να πετύχουμε του στόχου αυτού. Και υπάρχουν, ξέρετε, η ανισότητα, για παράδειγμα, παρά το γεγονό ότι είμαστε οι τρίτοι στον κατάλογο ισότητα στον κόσμο, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά στοιχεία που αυξάνουν την ανισότητα αν δεν υπάρχει συστηματική πολιτική καταπολέμηση της ε, ανισότητας. Και αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα. Τα προβλήματα της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, γιατί η μετανάστευση προφανώς προκαλεί ανισότητες, είναι πολύ πιο δύσκολο καταλαβαίνετε, να βρει κανεί δουλειά, εισόδημα, χωρίς να μιλάει τη γλώσσα, χωρίς να μιλάει, χωρίς να έχει το εκπαιδευτικό υπόβαθρο το οποίο κατανοούμε εμείς. Και αυτό επηρεάζει αφορά και την ε, συμμετοχή στην αγορά εργασία. Ελπίζω λοιπόν και φαντάζομαι ότι όλες οι χώρες θα το κάνουν αυτό. Η Πρόεδρος ε, αναρωτιέμαι αν ρωτούσαμε στο Συμβούλιο πόσες χώρες το κάνουν αυτό, γιατί σε πολλές χώρες ε, αυτή η στόχη φαίνεται ότι αποτελούν αναπτυξιακό ζήτημα και ήμασταν εδώ με την Επιτροπή Περιβάλλοντος σήμερα το πρωί γιατί συνεργάζονται οι δύο, οι δύο επιτροπές μας. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει αρκετή συνείδηση για το θέμα αυτό, γιατί ξέρουμε τους, ε, ότι υπάρχουν αυτοί οι βιώσιμοι αναπτυξιακοί στόχοι. Είναι πολύ εντυπωσιακά αυτά που μας είπατε για την κατανομή των στόχων ανά Υπουργείο. Και φαντάζομαι ότι αν ρωτούσαμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιο είναι ο αρμόδιο αναγενική διεύθυνση για τον κάθε στόχο, ούτε αυτοί θα ήξεραν. Συνάδελφοι, θέλετε να πάρετε το λόγο να θέσετε ερωτήσει ε, προ την ε, Υπουργό, προ την Πρωθυπουργό, η κυρία Φαμπρέμπτ. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει πρώτα απ' όλα να σα πω ότι είναι μεγάλη η τιμή μα ε, που σα έχουμε μαζί μα και νομίζω ότι δεν πρέπει να είσαστε πολύ μετριόφρον γιατί γνωρίζουμε ότι η Νορβηγία είναι από τις πιο προχωρημένες χώρες σε όλα τα επίπεδα της ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, γι' αυτό λοιπόν ε, εντάξει, καταλαβαίνω ότι μπορεί και εσείς να θέλετε ε, να έχετε σχέδια για να βελτιωθείτε όλο και περισσότερο, αλλά παρόλα αυτά σε σχέση με άλλες χώρες είστε πολύ μπροστά το θέμα της ψυχικής ε, και πνευματικής υγείας ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε και εμείς ε, το ίδιο πρόβλημα. Και εμείς πρέπει να πω ότι δεν έχουμε τόσο πολύ ανισότητα. Είναι η ευημερία αρκετή σε αρκετά μεγάλο βαθμό στη χώρα μου το Βέλγιο, αλλά παρόλα αυτά έχουμε πρόβλημα όσον αφορά την ψυχική υγεία. Επίσης, τα ζητήματα διακυβέρνησης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η Λίντα ήδη αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Ε, ένα από τα θέματα που με προβληματίζουν και με απασχολούν είναι το εξής. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ε, αυτά που λέμε δεν παραμένουν σε επίπεδο καλών προθέσεων ε, και ότι, ε, εν πάση περιπτώσει, θα υπάρξει υλοποίηση. Έχουμε μία μεθοδολογία, έχουμε ένα τρόπο εργασίας για το πώς μπορούν κάποια πράγματα να υλοποιηθούν στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτά τα ζητήματα πρώτα απ' όλα εν το οίκο μας. Δηλαδή, προγράμματα και ωραία λόγια έχουμε. Το ζήτημα είναι ότι εξακολουθούμε να έχουμε πολλά προβλήματα διακυβέρνηση. Ακόμα και στα πλαίσια τη Κομισιόν υπάρχουν ένα σωρό ε, μονάδες διοικητικές, ε, γενικές διευθύνσει κλπ. που ασχολούνται με τα ίδια θέματα. πώ μπορεί να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά τη ε, διακυβέρνηση. Επίση, αν εσεί είσαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα λέγατε, τι θα προτείνατε. Να υπάρχει ένα επίτροπο του οποίου το χαρτοφυλάκιο θα είναι ακριβώ αυτό, η καλύτερη διακυβέρνηση. Πώ μπορούμε να επιτύχουμε λοιπόν υλοποίηση των στόχων εντό Ευρωπαϊκής Ενώσεω. Πρόεδρος, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο, θέλουν να υποβάλουν κάποιο ερώτημα στον Πρωθυπουργό. Όχι. Να απαντήσει λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι ένα, μία από τις προκλήσεις οπωσδήποτε είναι ότι κάποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ε, βρίσκονται εκτός αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας πούμε η εκπαίδευση, οι υπηρεσίες υγείας, ε, είναι εκτός ε, των αρμοδιοτήτων και επομένως ε, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αλληλοκάλυψη αυτών των θεμάτων. Υπάρχουν ζητήματα όμως επί των οποίων όντως υπάρχει η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν και οι αντίστοιχοι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Επομένως αυτό θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε καλά αυτούς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που εμπίπτουν σε αρμοδιότητες και επομένως να γίνει η απαραίτητη προσαρμογή. Ε, ε, και αυτό που είπατε ε, τα τελευταία 15 χρόνια αρκετά καλά τα πήγαμε εγώ που τα βλέπω και απ' έξω ναι αρκετά καλά αλλά νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα, αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να τα θέσετε σε όλες τις μεθοδολογίες που ακολουθείτε και τις πράξεις που ακολουθείτε. Ας πούμε τρομοκρατία. Πώς αντιμετωπίζετε το ζήτημα της τροποκρατίας, πώς εντάσσετε την κοινωνία των πολιτών μέσα σε αυτό το ζήτημα. Γιατί ναι, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ε, έρχονται με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο και ενδεχομένως δεν μπορούν να προσαρμοστούν καλά ή αισθάνονται ε, ότι ε, δεν εντάσσονται καλά στην κοινωνία Νομίζω ότι μπορείτε να ε, εφαρμόσετε πιο συμπεριληπτικές ε, πολιτικές έτσι ώστε ε, μέσα να συμμετέχουν οι άνθρωποι αυτοί σε ομάδες νέων και σε άλλες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών ώστε να εντάσσονται καλύτερα. Το ζήτημα δεν είναι ε, να τα βάλουμε όλα σε έναν άβακα και να πούμε αυτό ισχύει, το άλλο το έχουμε κάνει καλά ή όχι. Ε, η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ε, και η απασχόληση των νέων οπωσδήποτε περνάει μέσα από τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης γιατί ακριβώς αυτοί οι στόχοι έχουν σαν κύριο σκοπό το να δώσουν ελπίδα ε, στις ε, επόμενες γενιές. Επομένως, ε, διασταύρωση των προσόντων και τέριασμα των προσόντων με τις προσπάθειες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτά είναι μικρά βήματα, πολύ σημαντικά. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ανταποκριθεί σε όλους τους στόχους. Μπορεί όμως να ανταποκριθεί στον υπαριθμό 16 που είναι η καλή διακυβέρνηση που αφορά την διαφάνεια, που αφορά τον σεβασμό της κοινωνίας των πολιτών. Ε, αυτά είναι ζητήματα τα οποία βρίσκονται υποπίεση σε πολλές χώρες ε, την σήμερα ημέρα. Επίσης, ε, στον στόχο 16 συμπεριλαμβάνεται και η διαφθορά. Υπάρχουν οι πόροι οι οποίοι μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα να λυθούν αυτά τα κοινωνικά ε, προβλήματα και προβλήματα όπως είναι η διαφάνεια ή η διαφθορά. Αυτά θα πρέπει, εκεί θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, δυστυχώς δεν έχουν ξεφύγει ακόμα από την, ε, από την κίνηση ε, οι ομιλητές μας. Θα δώσω λοιπόν το λόγο σε συνάδελφο Νταλή. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πρωθυπουργέ που ήρθατε εδώ Σας άκουσα με μεγάλη προσοχή να αναφέρεστε κυρίως στην ε, ψυχική ε, υγεία ε, και με μεγάλη χαρά σας άκουσα να το αναφέρετε αυτό γιατί δυστυχώς πολύ συχνά δεν περιλαμβάνεται στους πολιτικούς στόχους σε πολλές χώρες και εσείς τον περιλάβατε και είναι πάρα πολύ θετικό. Είπατε ότι έχετε καταγεγραμμένες 500 αυτοκτονίες αναέτο, Εγώ όμως πιστεύω ότι αυτή είναι μονάχα η κορφή του παγόβουνου, γιατί όταν μιλάμε γενικότερα για την ε, πνευματική ψυχική υγεία, ε, οι άνθρωποι που τους αφορά το ζήτημα είναι πολύ περισσότεροι. Επίσης αναφερθήκατε ε, στην εκπαίδευση και αναφερθήκατε και στην μετανάστευση ζήτημα ζέων για την ώρα. Είναι ζητήματα τα οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Εσείς στη χώρα σας πώς βάζετε τις προτεραιότητες σε σχέση με την ε, πνευματική υγεία, πώς την εντάσσετε δηλαδή αυτή την υγεία στις γενικότερες ε, ε, στο γενικότερο πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας. Επίσης, και για τα υπόλοιπα ζητήματα, πώς το διασυνδέεται. Δεύτερο, όσον αφορά δηλαδή τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ε, οπωσδήποτε ε, το κλίμα και η κλιματική αλλαγή αυτόματα γίνεται ε, προτεραιότητα. Ε, θα ήθελα να μας πείτε ίσως και κάποια λόγια σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την Συμφωνία των Παρισίων ε, και επίσης τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ξεπεράσουμε και αυτές τις συμφωνίες. Ποιες πιστεύετε ότι ε, μπορείτε να αντιμετωπίσετε συγκεκριμένες πολιτικές όπως είναι ας πούμε ε, η εμπορία ρήπων, όπως είναι τέτοιου είδους εμπορικές συμφωνίες πώς διασυνδέεται όλα αυτά τα ζητήματα. Να ξεκινήσω από την πνευματική υγεία. Είναι προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου. Η πνευματική υγεία και η σχέση της με την ε, κατάχρηση ουσιών, διότι ε, η τοξικομανία ή η κατάχρηση αλκοόλ συνδέεται με τα θέματα αυτά λέμε ότι όλα τα νοσοκομεία μας πρέπει να έχουν το ίδιο δυναμικό σε αυτούς τους τομείς που έχουν και για την ε, κανονική γιατρική. Η ε, νοσοκομιακή περίθαλψη είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης ε, στην Νορβηγία. Έτσι λοιπόν έχουμε πολλή επιρροή. Είπαμε λοιπόν ότι θα αξιολογήσουμε την ηγεσία των νοσοκομείων ανάλογα με το αν μπορούν να δείξουν ότι έχουν αυξήσει τις δαπάνες για την πνευματική υγεία και για, ε, την, για, για, την κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών ε, περισσότερο από ό,τι έχουν αυξήσει τις ε, άλλες τους δαπάνες. Αυτό είναι το ένα που κάναμε. Το άλλο είναι ότι σε συνεργασία με τους Δήμους ε, ασχολούμαστε με τη δουλειά εκτός νοσοκομείων. Αυτό όμως είναι λίγο πιο δύσκολο, διότι και οι Δήμοι έχουν κάποια ανεξαρτησία. Έχουμε όμως σχέδιο δράσης για την τοξικομανία. και οι ανθρώπους που βρίσκονται σε περίοδο αποκατάστασης. Αυξάνουμε τις επιδοτήσεις για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε εργασία και στέγαση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην ξαναπέσουν στην ε, κατάχρηση ουσιών. και μαζί με τα κόμματα που μας στηρίζουν στο Κοινοβούλιο εκπονούμε ένα σχέδιο δράσης για τα προβλήματα υγείας των νέων. Διότι διαπιστώνουμε ότι αυτά αυξάνονται. Θα έχουμε λοιπόν ένα ειδικό σχέδιο δράσης με δικούς του πόρους και ξεκινήσαμε αυξάνοντας τις υπηρεσίες υγείας στα σχολεία οι νοσοκόμες στα σχολεία δηλαδή, Έχουμε νοσοκόμες στα σχολεία, έχουμε και ψυχολογική βοήθεια μέσω των Δήμων. Είναι όμως πράγματα που πρέπει να κάνει κανείς και στα οποία πρέπει να δώσει προτεραιότητα. Ε, η ασθένεια που είναι πιο πιθανό να πλήξει κάποιον ε, στην Νορβηγία είναι οι διανοητικές παθήσεις ε, και, ε, και εάν δεν λάβει κανείς ε, εγκαίρως βοήθεια μπορεί να χειροτερέψει πολύ η κατάσταση και μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι αυτό συμβαίνει επειδή ζούμε σε δύσκολους καιρούς, επειδή είναι πιο προηγμένες οι κοινωνίες μας, επειδή συναντάει κανείς προβλήματα στην καθημερινή του ζωή, στην εργασιακή του ζωή. Και ίσως κάποιοι να θεωρήσουν ότι δεν πρέπει να δώσουμε τόση σημασία στις ψυχικές ασθένειες, διότι ε, τότε απαιτούνται και περισσότεροι πόροι για αυτές τις ασθένειες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα. Το δεύτερο θέμα που αναφέρατε ήταν η αλλαγή του κλίματος. Ε, εγώ είμαι υποστηρίκτρια της ε, Συμφωνίας του Παρισιού. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με βάση αυτήν. Να πούμε ότι εντάξει, οι Ηνωμένε Πολιτείε αποφάσισαν να ε, αποσυρθούν, αλλά οι υπόλοιποι θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω στο θέμα αυτό και νομίζω ότι θα μας εκπλήξει το πόσα θα κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείες παρά την ηγεσία τους. Ήδη βλέπουμε χαμηλότερες εκπομπές και νομίζω ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Εμεί εργαζόμαστε πάνω στο δικό μας σχέδιο να μειώσουμε τι εκπομπέ ε, κατά 40%. Νομίζω ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών γίνεται πιο σφιχτό. Πρέπει να ανέβει η τιμή του διοξιδίου του άνθρακα για να πετύχει κανείς τα αποτελέσματα που θέλει μέσω του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Στον τομέα εκτός συστήματος εμπορίας εκπομπών, Ε, θέλουμε να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στις, ε, στα μέσα μαζικής ε, μεταφοράς. Διότι ο τομέας αυτός αντιπροσωπεύει μεγάλο ποσοστό. Διότι εμάς το ρεύμα μας παράγεται κυρίως με υδροελεκτρικά εργοστάσια. Οι μεταφορές όμως είναι σημαντικός τομέας. Επίσης, οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να τρώνε κόκκινο κρέας. Ε, μπορούμε να τους ενθαρρύνουμε να τρώνε λιγότερο, αλλά δεν γίνεται κανείς πολύ δημοφιλής ως πολιτικός αν ε, κουνάει το δάχτυλο και λέει ότι πρέπει να τρώτε λιγότερο κόκκινο κρέας. Γι' αυτό αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε στο τομέα των μεταφορών. Σήμερα, στην Ορβηγία, τα νέα οχήματα είναι ηλεκτρικά και έχουμε πολύ χαμηλή φορολογία τα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Ε, προσπαθούμε με τέτοια φορολογικά κίνητρα να αλλάξουμε την συμπεριφορά των ανθρώπων. Θα είναι όμως δύσκολο να πετύχουμε μείωση κατά 40% στον τομέα εκτός συστήματος εμπορίας εκπομπών. Πιστεύουμε όμως ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας μέχρι το 2030. Ήδη τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλύτερα από ό,τι νομίζαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η τη Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που βλέπω εδώ Πρωθυπουργό ε, από μία από τις βόρειες χώρες εδώ στην ε, αίθουσά μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την ε, ανθρωπιστική βοήθεια και συνεργασία. Θαυμάζω πολύ αυτά που κάνει η Νορβηγία στον τομέα αυτών. Τι προτείνετε εσείς όσον αφορά την χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς επίτευξη των στόχων ε, της χιλιετίας. Βλέπω μια ε, αρκετά ανησυχητική εξέλιξη να συνδέει κανείς ε, την ανθρωπιστική βοήθεια με τον έλεγχο της μετανάστευσης στην Ευρώπη. Ναι, κατά τις διαπραγματεύσεις μας ε, αυτό ήταν ε, πολύ σημαντικό θέμα για το Κοινοβούλιο. Θέλαμε να αντιμετωπίσουμε την ε, φτώχεια. Η κυρία Σόλμπεργκ, ναι, είναι πολύ δύσκολα τα θέματα αυτά. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι σε κάποιους τομείς, εάν δεν καταφέρουμε να έχουμε έλεγχο της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια, δεν θα μπορέσουμε να προσφέρουμε βοήθεια στους ανθρώπους. βλέπω να θίγονται θέματα ασφάλειας και στο θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Θέλουμε να, να φτάσουμε στους πιο ευάλωτους ε, ανθρώπους. Ουσιαστικά μια σύνοψη των ε, στόχων είναι να μην αφήσουμε ε, κανέναν πίσω. Εγώ πιστεύω ότι η ανάπτυξη ποτέ δεν μπορεί να ε, επιβληθεί απ' έξω. Αναπτύσσεται εντός μιας χώρας μέσω της πολιτικής που ε, ενθαρρύνει την ανάπτυξη. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε. Εάν στηρίζουμε πολιτικούς και συστήματα με θεματολόγιο ανάπτυξης στο οποίο πιστεύουμε, μπορούμε να το στηρίξουμε ή μπορούμε να, ε, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους ε, όταν αντιμετωπίζουν φτώχεια. Μπορούμε να στηρίξουμε την εκπαίδευση, διότι εάν εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους, θα μπορούν οι ίδιοι να επιφέρουν την αλλαγή. Θα πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια μερικές φορές ε, στηρίζει συστήματα που δεν ε, στηρίζουν την ανάπτυξη. Πάντα υπάρχει αυτή η πτυχή. Ο συμπρόεδρος μου, που δεν είναι παρόν σήμερα, ο πρόεδρος της Γκάνας, έχει πει ότι η φιλοδοξία θα πρέπει να είναι, να είναι κανείς ανεξάρτητος από την ανθρωπιστική βοήθεια και είναι πολύ καλός αυτός ο στόχος. Διότι σε πολλές χώρες, εάν υπάρχει διαφάνεια, υπάρχουν πόροι και το βλέπουμε αυτό ε, και στις χώρες όπου υπάρχει πολλή διαφθορά. Υπάρχουν ε, χρήματα. Βλέπω ότι καταφτάνουν οι φίλοι μου ε, από τους υπερασπιστές των στόχων της χιλιετίας. Μπορεί να έχουν διαφορετική θέση, αλλά η βοήθεια θα οδηγήσει σε ανάπτυξη μόνο εάν υπάρχει κυβέρνηση, εάν υπάρχει ένα σύστημα που πιστεύει στην αναπτυξιακή πολιτική. Τότε μπορεί κανείς να επενδύσει στην υγεία και στην εκπαίδευση, διότι έτσι επενδύει στους ανθρώπους. Δεν θα μπορέσουμε όμως να έχουμε ανάπτυξη εάν δεν βοηθάει το σύστημα. Κύριε Πρωθυπουργέ, μας δείξατε γιατί επέλεξαν εσάς ως συμπρόεδρο να ευχαριστήσουμε την ε, Πρωθυπουργό που μας έδειξε έτσι με αυτοσχέδιο τρόπο πόσο έχει συμβάλει η χώρα της στην επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Well, our guests have been on a kind of odyssey. Φαντάζομαι ότι είχατε περιπέτειες στις Βρυξέλλες. Οδύσσια ολόκληρη. Γι' αυτό σας πήρε τόσο χρόνο που να φτάσατε, μέχρι να φτάσατε. Χαιρόμαστε ωστόσο που καταφτάσατε και να ενημερώσω τους προσκεκλημένους μας ότι συζητούσαμε πριν από την αφήξή σας για τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Είδαμε ένα σύντομο βίντεο, συζητήσαμε για το πώς ε, σήμερα το πρωί την Ευρωπαϊκή ημέρα ανάπτυξης ε, υπογράψαμε μια νέα συνένεση για την ανάπτυξη και την ένταξη στο νομοθετικό σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα πλαίσιο συνεργασίας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι λοιπόν γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό σας στάση. Ιδιαίτερα σήμερα σε μια εποχή που η πολυμέρεια, η πολυμερή συνεργασία μα υπονομεύεται. Ήμουν στην Κοπενχάγη και πραγματικά ήμουν πολύ απογοητευμένη. Μετά πήγαμε στο Παρίσι, μείναμε ικανοποιημένοι. Τώρα κάνει πίσω η ηγεσία της Αμερικής. Ελπίζουμε ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει στην εφαρμογή και υλοποίηση των στόχων της Συμφωνίας του Παρισίου και σε ό,τι αφορά τους στόχους, τους βιώσιμους. Θα πρέπει πλέον να γίνουν τα λόγια πράξη και να μην μείνουν κενά λόγια στον αέρα. Να μην καθυστερήσουμε, να ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη συζήτηση στο πρώτο πάνελ. Αν ο καθηγητής ε, Σάξ ε, είναι έτοιμο και κατάφερε να ξελαχανιάσει μετά από αυτή την Οδύσσια στις Βρυξέλλες. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν ε, από το Πανεπιστήμιο της Κολόμπια ο καθηγητής Τζέφρι Σάξ, ο οποίος έχει παρευρεθεί σε διάφορες περιστάσεις εδώ στο Κοινοβούλιο και προσβλέπουμε και ανυπομονούμε να ακούσουμε την παρουσίασή σας, ε, καθηγητή Σάξ. Ε, σας ευχαριστώ και μεγάλη τιμή και χαρά πάντα να βρίσκομαι μαζί σας. Ε. Η ατζέντα για τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους είναι εξαιρετικά σημαντική. Η ΕΠΑ θα κάνουν ένα διάλειμμα γιατί βρισκόμαστε σε μια αναφραγουμένου περίεργη πολιτική κατάσταση και πιστέψτε μου ότι εμείς από αυτή την πλευρά του Ατλαντικού θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την πολιτική κατάσταση, γιατί είναι πραγματικά ε, φρικτό, επικίνδυνο και απαράδεκτο ως κατάσταση. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά εν τω μεταξύ ο κόσμος θα πρέπει να κινηθεί προς το εμπρός προφανώς και η Ευρώπη. Προφανώ έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη Κοιτώντα που βρίσκονται οι χώρε σε ό,τι αφορά του βιώσιμου αναπτυξιακού στόχου, η Ευρώπη με μεγάλη διαφορά είναι η πιο προηγμένη ε, περιοχή στον κόσμο σε ό,τι αφορά την ατζέντα αυτή. Γιατί πιστεύω ότι άλλωστε ε, η ατζέντα αυτή αποτυπώνει τι ευρωπαϊκέ αρχέ και αξίε. Γιατί πρόκειται για μια περιοχή η οποία επιμακρών εστιάζεται στου τριπλού στόχου τη οικονομική ευημερία, κοινωνική συμπερίληψη και περιβαλλοντική αηφορία. Αλλά και στο εσωτερικό της Ευρώπης υπάρχουν κάποιες σημαντικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ο ρόλος δε της Ευρώπης ε, στον υπόλοιπο κόσμο είναι κρίσιμη σημασία και κυρία σημασία. Να πω δύο λόγια λοιπόν για όλα αυτά τα ζητήματα. Στο εσωτερικό τη Ευρώπη, η πιο σημαντική πρόκληση, θεωρώ, πέρα από τα καθημερινά ζητήματα διαχείριση τη οικονομία και ε, τη οικονομική ανάπτυξη των διαφορών χωρών με διαφορετικού ρυθμού. Το πιο σημαντικό ω ε, ως ευρωπαϊκή πρόκληση είναι η μετα... Είναι τα ενεργειακά συστήματα. Χρειάζονται λοιπόν ε, στόχοι. Χρειάζεται ένα σχέδιο για την επίτευξη των στόχων. Δεν μπορούμε να έχουμε 28 διαφορετικά εθνικά σχέδια όμως για την επίτευξη των στόχων. Χρειάζεται όμως ένα ενιαίο σύστημα. Θα πρέπει να μεταφέρεται η ενέργεια από το ένα μέρος στην Ευρώπη στο άλλο, στην άλλη άκρο της Ευρώπης. Ε, ηλιακή ενέργεια θα πρέπει να χρησιμοποιείται και στη Βόρεια Ευρώπη, γιατί στην παρούσα φάση δεν υπάρχει καν ενεργειακό πλέγμα που θα μπορούσε να βοηθήσει τη μεταφορά αυτή της ενέργειας. Ως τώρα, για τη μεταφορά και την ενεργειακά συστήματα θα έπρεπε να υπάρχει συμφωνία 28 διαφορετικών χωρών με 28 διαφορετικά εθνικά συστήματα και το ξέρω ότι είναι σκληρό αλλά χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό σχέδιο. Χρειάζεστε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο όπως και οι ΙΠΑ χρειάζονται να συνδέσουν τα τρία υποδικτυά τους για να υπάρχει ένα ενιαίο δικτύο, για να μην υπάρχει ε, τέτοιο κατακαιρματισμό. Και αν δεν υπήρχε αυτή η παράλογη πολιτική κατάσταση, θα συζητούσαμε πώ θα ενώσουμε του από την Ανατολική στη ακτή για να μεταφέρουν ε, ενέργεια σε όλες τις ΗΠΑ και πώ μπορεί να συνδεθεί η καναδική υδροελεκτρική ενέργεια με το βορείο-ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Χρειάζονται στρατηγικέ, λοιπόν, μία ενιαία στρατηγική η οποία θα καλύπτει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι το βασικό, αυτή είναι η βασική συμβουλή που έχω να σας δώσω. Να βρείτε ένα ευρωπαϊκό τεχνικά προηγμένο σχέδιο για να σας είναι σαφές που θα είναι οι γραμμές και τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας. Γιατί κάποιες χώρες είναι υπέρ της πυρηνικής ενέργειας, κάποιες άλλες κατά αλλά χρειάζεται ένα λες ανθεκτικό, αξιόπιστο σύστημα ενέργειας στην Ευρώπη, σε, το οποίο θα χρησιμοποιεί και άνθρακα. Το 2030 είναι ένα βήμα, ένα στόχο, το 2050 αποτελεί mm. ένα περαιτέρω στόχο. Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί τη βασική πρόκληση για την Ευρώπη σε ό,τι αφορά τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Άλλη μια πρόκληση η οποία συνδέεται με αυτή είναι η βιοπικιλία, η χρήση των γεών, η κρίση της Μεσογείου, η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρή και ως εκ τούτου οι βιώσιμοι αναπτυξιακοί στόχοι υπαριθμών 14 και 15 έχουν ιδιαίτερη ε, εφαρμογή εδώ. Πρόκειται για ένα υπέροχο τμήμα του πλανήτη, ακόμα και αν πολλές φορές έχουμε την αντίθετη αίσθηση. Πρόκειται για ένα πραγματικά πολύ εντυπωσιακό κομμάτι του κόσμου, το οποίο προσεγγίζει τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστούν τα περιβαλλοντικά, οι περιβαλλοντικοί στόχοι ε, με οργανωμένο, συντονισμένο τρόπο. Γίνεται, αλλά κατακριματισμένα δεν γίνεται ακόμα με οργανωμένο τρόπο, γιατί επικρατεί το εθνικό επίπεδο και όχι το ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι επαρκώς σε βάση περιπτώσει. Αυτή θα ήταν η βασική μου σύσταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης μάλλον, σε όλο τον κόσμο, θα έπρεπε να είναι πολύ πιο μεγάλος από ό,τι έω τώρα. Γιατί προφανώς στα συστήματα που εγκαθιδρύθηκαν μετά τον Δεύτερο Πόλεμο, έχουν πλέον εκπνεύσει, βρισκόμαστε σε ένα διαφορετικό, σε μια διαφορετική χρονική περίοδο. Έχουμε ένα πολιτικό πόλεμο στη ΣΥΠΑ, έναν εντελώς παράλογο πολιτικό πόλεμο, αλλά η ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιβιώσει χωρίς πολιτική εξωτερικών υποθέσεων, ότι εντάξει δεν πειράζει φτάνει και το ΝΑΤΟ, θεωρώ ότι πλέον είναι παροχημένη, γιατί η Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια έχει πέσει θύμα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και των προσφυγικών ροών. Δεν προήλθαν από το πουθενά οι πρόσφυγες από την εισβολή στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, από το μυστικό πόλεμο στη Συρία, με τη Σαουδική Αραβία, από τη ΣΥΠΑ, από την Γαλλία και τη ΣΥΠΑ που εισέβαλαν στην Λιβύη χρειάζεστε πραγματικά καλύτερη πολιτική εξωτερικών. Λυπάμαι λοιπόν, που σας το λέω, το λέω έξω από τα δόντια. Γιατί γι' αυτό αποσταθεροποιήθηκε η Ευρώπη. Πρόκειται για τον αντίκτυπο και την επιρροή της πολιτική των ΗΠΑ. Τώρα ξαφνικά οι ΗΠΑ μιλάνε για τον Ιράν. Πλάκα μα κάνετε. Δεν ε, μας φτάνουν αυτά που έχουμε καθημερινά. Αλλά έχουν ήδη τα τύμπανα του πολέμου, το οποίο είναι πραγματικά εντελώ παράλογο και πάρα πολύ επικίνδυνο. Μα πού είναι η Ευρώπη να σηκωθεί να πει σταματήστε πια, Σόνι, ω εδώ. Αυτό είναι, θεωρώ, ο ρόλο τη Ευρώπη. Πρόκειται για την πιο μεγάλη ενοποιημένη αγορά του κόσμου και θα πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ευρώπης με πιο συντονισμένο τρόπο, όχι μόνο μέσω της Δυτικής ε, Συμμαχίας, της Συμμαχίας των Δυτικών χωρών, με τους ε, περίεργους αυτούς εταίρους ε, της Αμερικής, που φαίνεται ότι αδιαφορούν τα θέματα αυτά. Πολύ φοβάμαι. Από πλευράς αξιών και ψυχολογικά, η Ευρώπη είναι ο φυσικός ηγέτης για όλα αυτά τα θέματα και θα πρέπει να έχει πιο έντονη παρουσία. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, οι βιώσιμοι αναπτυξιακοί στόχοι αποτελούν μια ευκαιρία για να επιληθούν προβλήματα, γιατί ουσιαστικά αποτελούν ένα παζλ, αν θέλετε. Ένα στόχο που είναι, για παράδειγμα, για, κρίσιμος για το μέλλον της Ευρώπης είναι ο υπαριθμό 4, που αναφέρει ότι η καθολική α, δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να ολοκληρώνεται. Γιατί είναι αυτό τόσο βασικό. Έχετε 1,2 δις ε, άτομα στην Αφρική τώρα και ο πληθυσμός της Αφρικής θα φτάσει 4 δισεκατομμύρια αν συνεχιστούν οι τρέχουσες ε, ε, τάσεις εκτός και αν κάθε, παιδί, κάθε κορίτσι λάβει σωστή δευτεροβαθμία εκπαίδευση. Αν δεν ε, πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος λοιπόν ο υπαριθμό 4 θα είναι δημογραφικά ε, μη βιώσιμη η Αφρική και η Ευρώπη. Άρα το παζλ είναι ακριβώς, ο γρίφος ακριβώς είναι το πώς θα πετύχουμε αυτόν τον στόχο υπαριθμών 4, το πώς θα μπορεί κάθε παιδί στην Αφρική να ολοκληρώνει τη δευτεροβόηθμη εκπαίδευση, όταν στην παρούσα φάση το ποσοστό αυτό είναι στο 25%. Άρα ο στόχος τι προβλέπει ότι σε 13 χρόνια θα πρέπει να πάει μέσα από το 25% στο 100% για τη συμπλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι αυτό εφικτό. Είναι. Είναι λέγω. Αν μπορεί κανείς 8 χρόνια να πάει και να έρθει από το φεγγάρι, μπορεί να βάλει και όλα τα παιδιά στο σχολείο. Χρειάζεται σχέδια για να το πετύχουμε. Έμα ε, βέβαια. Υπάρχει αυτό το σχέδιο. Όχι, δεν υπάρχει. Θα μπορούσαν οι αφρικανικές χώρες να το κάνουν αυτό μόνοι τους. Ούτε αυτό. Τα έχω βγάλει και τα έχω μετρήσει 20 φορές. Από την καλή και από την ανάποδη. Σε όλες μου τις θέσεις στο σύστημα του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση της Νορβηγίας χρηματοδότησε την Επιτροπή Μπράουν για την εκπαίδευση και είπαν ότι έχουμε ένα χάσμα 40 δισεκατομμυρίων, 14 δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο. Ποιο θα παίρνει όμω αυτό σοβαρά ότι έχουμε 14 εκατομμύρια που, δισεκατομμύρια που μα λείπουν και χρειάζονται αυτά τα 14 δισεκατομμύρια για να βγάλουμε ένα εθνικό σχέδιο για την εκπαίδευση. Κανένα. Μηδέν άτομα. Τι κάνουμε λοιπόν για να κατανοήσουμε, να βγάλουμε ένα προπολογισμό, να εκτιμήσουμε τη σημασία των στόχων και τελικά όμω δεν καταρτίζεται κανένα σχέδιο για την επιτεύξη των στόχων αυτών. Οπότε εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξή που ήταν πολύ πιο φτηνό να πετύχουμε και να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε τους στόχους αυτούς από το να τους συζητάμε συνέχεια. Γιατί αν δεν πετύχουμε τους στόχους αυτούς, θα είναι τεράστιες και φρικτές οι συνέπειες και ήδη συμβαίνουν και θα χειροτερεύσουν, θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Αν υπήρχε ένας υπουργός ε, Εκπαίδευση παιδεία για την ε, Ευρώπη και την Αφρική και έλεγε ότι έχουμε πρόβλημα χρηματοδότησης, μα λείπουν κονδύλια, πώς θα το καλύψουμε, θα υπήρχε κάποιο σχέδιο, αλλά ό,τι πιο κοντινό πιστεύω ότι υπάρχει είναι η Επιτροπή μαζί με την Αφρικανική Επιτροπή. Θα έπρεπε να τα βάλουν κάτω και να πούν ότι κοιτάξτε, ξέρουμε πλέον ότι για να πετύχουμε τον αναπτυξιακό στόχο υπερθμό 4 ε, είναι βαρύ είναι βαριέ οι συνέπειε και θα πρέπει να τα πετύχουμε όλα αυτά. Δίνει πολύ βοήθεια η Ευρώπη, αλλά όχι στοχευμένα για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματο. Άρα, η σύστασή μου και πραγματικά αποτελεί μια συμβουλή και μόνο είναι να πάρετε το στόχο αυτό στα σοβαρά. Να ρωτήσετε και να ζητήσετε από τους επιτρόπους να σας πούν πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι ε, χώρε τη άμεση γειτονιά σα, ε, ποιο θα πρέπει να είναι ο ρόλος μας, ποια είναι τα κενά που υπάρχουν και πώ μπορούν να καλυφθούν τα κενά αυτά. Και θα κλείσω λέγοντα ε, ένα πράγμα, κάνοντα μια παρατήρηση η οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρη στην παρούσα φάση. Και χρησιμοποίησα και προηγουμένω το παράδειγμα αυτό και ζητώ συγγνώμη από του συναδέλφου που το ξανακούν, ο Κέννεντι, ο πρόεδρος Κέννεντι το 61. Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα για το φεγγάρι, για το ταξίδι στο φεγγάρι, δεν είπε ότι «Α, πιστεύω ότι θα ήταν εξαιρετικό να ε, κατατήσουμε ένα πρόγραμμα για το διάστημα». Δεν είπε «Τι ωραίο το φεγγάρι, Μ, πολύ ενδιαφέρον θα ήταν να το επισκεφτούμε». Ούτε είπε «Δεν πάμε στο φεγγάρι και να ξαναγυρίσουμε με ασφάλεια». Όχι. Αυτό που είπε κατά λέξη ήταν πριν τελειώσει η δεκαετία αυτή να στείλουμε έναν άνθρωπο στο φεγγάρι και να επιστρέψει μετά στη γη. Έδωσε τον στόχο, έδωσε και το χρονικό πλαίσιο. Και ότι μετά τα πάντησαν πάρα πολλά χρήματα. Έβαλαν 500.000 άτομα στην NASA και 20.000 εταιρείε οι οποίες εμπλέκονταν και μετά μέσα σε 8 χρόνια ο Νίλ Άρμστρομ βρέθηκε να περπατάει στο φεγγάρι. Αυτό σημαίνει προγραμματισμός βάσει σχεδίου. Υπάρχει χρονικό πλαίσιο, υπάρχει στόχος και υπάρχει και μία σειρά βημάτων για να επιτευχθεί και η NASA ήταν ε, η πιο ιδιόρυθμη, θέλετε, σχετική υπηρεσία στον κόσμο. Ένα σωρό μηχανικοί οι οποίοι βγήκαν και είπαν ότι αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θέλουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο. Έχουμε λοιπόν ένα χρονοδιάγραμμα για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για την υγειονομική περίθαλψη. Έχουμε το χρονοδιάγραμμα, όχι αυτό που αποφασίσαμε εμείς, αυτό που μας ε, υπαγορεύει η φύση για την ε, μείωση των εκπομπών άνθρακα και για την ε, χρήση του άνθρακα. Τόσος μας μένει. Η ελπίδα μου και η έκκληση που απελαμβάνω κάθε μέρα δεκάδες φορές είναι Ας πάρουμε πια στα σοβαρά του στόχους μα αυτού, προκειμένου να έχουμε το χρονοδιάγραμμα, να ξέρουμε τι χρειάζεται να χρηματοδοτήσουμε και να περάσουμε στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας. Αν το κάναμε αυτό, ο κόσμος πραγματικά θα ήταν πολύ όμορφο μέρος να ζει κανεί πιο ασφαλή, πιο αιθαλή και βιώσιμο, πολύ πιο ειρηνικό, πολύ πιο παραγωγικό. Αν πάρουμε στα σοβαρά του στόχου αυτού. Σα ευχαριστώ πολύ. Um, thank, thank, Άκουσα στο BBC ότι η UNESCO λέει ότι οι επενδύσεις στην εκπαίδευση στην Αφρική ε, έχει πέσει κατά 4% σε σχέση με πέρσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι επικεφαλής των προσπαθειών. Και τώρα που η χώρα μου αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι καλό θα είναι να δώσω την Προεδρία στον συναδελφό μου, τον Παύλ Πόκ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ήσουν μέντοράς μου κατά την πρώτη μου θητεία, ε, διότι Είμαστε σχετικά νέο κράτο. Είπατε βέβαια ότι ε, αυτό μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε λάθη, όπως και να έχει. Είμαι αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΕΝΒΗ και γι' αυτό θα... Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ε, είναι ουσιαστικά το ψωμοτήρι μας. Απέχουμε πολύ από το να πετύχουμε τους στόχους. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τους υπερασπιστές ε, των στόχων αυτών περισσότερο από ποτέ, τώρα που αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις προκλήσεις. Και δεν ε, αναφερθήκατε σε δύο από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, που είναι αφενός η αναλογικότητα, κάτι που δεν έχουμε πετύχει ακόμα, και επίσης να είμαστε συνεπείς. Διότι δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να επιδείξουμε συνέπεια. Δεν θυμάμαι ποιος είπε ότι οι Βρυξέλλες ε, είναι κόλαση, αλλά ε, σήμερα προφανώς οι ε, προσκεκλημένοι μας είχαν κολλήσει στην κίνηση. Όπως και να έχει, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον καθηγητή Μουχάμαντ Ιούνους που είναι ιδρυτής της Τράπεζας Κρέμιν και που είχε ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα μικροχρηματοδότησης. είναι ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες ε, της εποχής μας. Ε, το 2006 και η τράπεζα ε, Γκρέμιν και ο καθηγητής Γιούνους έλαβαν από κοινού το βραβείο Νόμπελ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Πολύ σύντομα θα σας μιλήσω για τη δουλειά που έχω κάνει και τη σχέση της με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Καταρχάς, έχω την τράπεζα ε, την οποία ίδρυσα πριν περίπου 40 χρόνια, μια τράπεζα που ε, δανείζει σε φτωχούς. Ε, σήμερα στο Παγκλατές έχουμε πάνω από 9 εκατομμύρια δανειστές, κυρίως γυναίκες. Δεν λαμβάνουμε δάνεια από άλλους οι χορηγίες. Έχουν έχουμε αρκετά κέρδη ώστε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε και τα κέρδη ε, πάνε στους ε, δανειστές που είναι και μέτοχοι. Αυτή λοιπόν είναι η μικροοικονομία, η μικροχρηματοδότηση. Πριν 9 χρόνια, το 2008, Ε, ξεκινήσαμε το ίδιο πρόγραμμα στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, είχαμε λοιπόν την Τράπεζα γραμμή ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε. 20 υποκαταστήματα έχουμε τώρα πια στις Ηνωμένε Πολιτείε, 8 στη Νέα Υόρκη μόνο, στο Λος Άντζελος, στο Σαν Φρανσίσκο και αλλού. 86.000 και κυρίως γυναίκες ε, έχουν ε, πάρει δάνεια από μας. Και στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ε, έγγραφα δικαιολογητικά να μας δώσουν. Όσον αφορά την απόδοση, όμως έχουμε δει εκπληκτικά αποτελέσματα. Συνεχίζεται λοιπόν το πρόγραμμα αυτό. Αυτό που θέλω να πω εδώ πέρα όμως είναι ότι είναι ότι εκτός από το Μπαγκλαντές μου έχει ζητηθεί από άλλες χώρες να δημιουργηθεί νομοθεσία για να δημιουργηθεί τράπεζα για τους φτωχούς. Η νομοθεσία για τις τράπεζες επιτρέπει τη δημιουργία τράπεζας για τους πλούσιους, αλλά χρειάζεται κανείς ξεχωριστό τραπεζικό σύστημα για τους φτωχούς. Γι' αυτό σας καλώ να εξετάσετε το θέμα αυτό. Στι Ηνωμένε Πολιτείε δανείζουμε χρήματα ω μη κυβερνητική οργάνωση. Δεν έχουμε άδεια λειτουργία τράπεζα. Εάν είχαμε άδεια λειτουργία σε τράπεζα, θα μπορούσαμε να φτάσουμε εκατομμύρια ανθρώπους. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει κανείς είναι να εγγυηθεί για να πάρει ο φτωχός ένα δάνειο. Η δεύτερη γενιά των δανειοληπτών μας ε, ε, έχουν λάβει πια εκπαίδευση. Έχουμε δώσει χρήματα για να πάνε σχολείο. Ε, δεν έχουν όμως εργασία. Ο άνθρωπος όμως ουσιαστικά είναι επιχειρηματίας. Σκεφτείτε τη μητέρα σας. Έχουμε μία μητέρα η οποία πήρε δάνειο, δεν έχει φύγει ποτέ εκτός του χωριού της, έγινε επιχειρηματίας. Εάν λοιπόν ε, έγινε η μητέρα σας, λέμε, σε αυτούς τους νέους ανθρώπους επιχειρηματίας, ε, πόσο μάλλον εσείς που ε, έχετε πάρει και κάποια εκπαίδευση. Σκεφτείτε λοιπόν καινοτόμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που έχω αναφέρει, ότι η ανεργία είναι τεχνητό πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι η απασχόληση, είναι η επιχειρηματικότητα. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε ένα κοινωνικό ταμείο επιχειρήσεων. Ζητάμε από τους νέους να μας υποβάλουν νέες ιδέες όπως έκαναν και οι μητέρες τους και ουσιαστικά συμμετέχουμε ως επιχειρηματίες, τους χρηματοδοτούμε και όταν τελικά έχουν επιτυχία, επιστρέφουν τα χρήματα που πήραν και μετά ε, μπορούν να ανεξαρτητοποιηθούν. Το μόνο που ζητάμε δηλαδή είναι τα χρήματα που έχουμε επενδύσει εμείς στην επιχείρησή τους. Με αυτή την ιδέα λοιπόν απλά δίνουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους και μέσω του συστήματος εκπαίδευσης ε, θέλουμε να πούμε στους ανθρώπους ότι ή θα αναζητείτε εργασία ή θα δημιουργήσετε θέσεις απασχόλησης. αλλά ουσιαστικά γεννηθήκατε για να δημιουργήσετε θέσεις απασχόλησης. Έχετε γεννηθεί ε, με αυτήν την ικανότητα δημιουργίας. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε μάθει να λύνουμε προβλήματα, γεωργοί, κυνηγοί, ε, συλλέκτες. Αυτή λοιπόν είναι η νοοτροπία που προσπαθούμε να εμφυτεύσουμε στους νέους. Κάτι που με ανησυχεί και που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, παρά όλα αυτά που σας είπα, είναι ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα συγκέντρωσης του πλούτου. Όλος ο πλούτος του κόσμου είναι συγκεντρωμένος σε λίγα χέρια. Είναι σαν ένα τεράστιο μπαλόνι με το κορδόνι. Το μπαλόνι λοιπόν μεγαλώνει συνεχώς. Το 99% του πλούτου όλου του κόσμου ανήκει στο 1% του πληθυσμού και η κατάσταση επιδεινώνεται. Το μπαλόνι φουσκώνει όλο και περισσότερο. Του χρόνου θα ακούσετε ότι περισσότερο από το 99% του πλούτου του κόσμου ανήκει σε λιγότερο από το 1%. Αυτός λοιπόν είναι ο κίνδυνος. Και αυτό οφείλεται στην τομή που έχουμε δημιουργήσει θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, διότι αλλιώς ε, θα είναι εκρηκτικό το θέμα, θα είναι μια ορολογιακή βόμβα. Ακούσατε κατά τη διάρκεια των εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο Μπέρνι Σάντερς έλεγε ότι το 1 δέκατο του ενό στα 100 του πληθυσμού κατέχουν παραπάνω από το 90% του πλούτου των Ηνωμένων Πολιτειών μία οικογένεια στις Ηνωμένε Πολιτείε, η οικογένεια που έχει την επιχείρηση Walmart, έχουν ε, τα περισσότερα χρήματα. Το πρόβλημα επιδεινώνεται κάθε χρόνο και δεν περιορίζεται στις Ηνωμένε Πολιτείε. Σε κάθε χώρο βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Όλο ο πλούτο βρίσκεται σε ελάχιστα χέρια. Ό,τι και να κάνουμε, αυτό θα συνεχίσει να χειροτερεύει και η κατάσταση θα γίνει πολιτικά εκρηκτική εκτό εάν ενεργήσουμε. Και το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι ε, στόχοι μας θα πρέπει να είναι τρία μηδενικά. Μηδενική φτώχεια, μηδενική ανεργία. Επειδή είναι τεχνητή έννοια μπορούμε να την εξαλείψουμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο επιχειρηματικότητας ώστε να μην χρειάζεται κανένας να παραμένει άεργος. Δεν έχει νόημα αυτό άλλωστε. Ε, όταν ε, ζούσαμε στα σπήλαια, ε, ένας άνθρωπος που δεν εργαζόταν ε, θα πέθαινε. Έπρεπε να βγει, να κυνηγήσει, να καλλιεργήσει. Αλλά το οικονομικό μας σύστημα δεν το ενθαρρύνει αυτό. Το θέμα είναι ότι αν βάλει κάποιο χρήματα στο τραπέζι, ο καθένας μας θα γίνει επιχειρηματίας. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε κόσμο με μηδενική ανεργία και το τρίτο μηδενικό που πρέπει να πετύχουμε είναι οι μηδενικές εκπομπές. Οι εκπομπές. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά για όσα μας είπατε. Έχουμε μπροστά μας ε, μεγάλα πράγματα. Έχουμε το, τη γη, έχουμε πλανήτες, έχουμε τη Unilever όπως ε, έλεγε και κάποιος. Εν πάση περιπτώσει, Έχουμε τώρα τον επόμενο μιλητή μας, ο οποίος είναι πρόεδρος ε, του Business Council ε, για τους ε, βιώσιμους στόχους ανάπτυξης. Επίσης είναι μέλος του Global Contact Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών και επίσης έχει ζητηθεί από, τις, από το, του ζητήθηκε από το Γενικό γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών να γίνει μέλος του Advocacy Group για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Σας δίνω μέσα στο λόγο κύριε κύριε ε, Πόλμαν. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά ακούω πάντα και ευχαρίστηση τον Τζέφρι και τον Μοχάμαντ όταν μιλάνε και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω ε, για τους στόχους αυτούς ο Γενικός ε, ε, Γραμματέας είχε μιλήσει ενώπιον των 27 τότε ε, μελών για να συζητήσει για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και είχε πει ότι αν δεν υπάρχει αξιοπρεπής συνολική διακυβέρνηση αυτό θα οδηγήσει σε πολύ μεγάλα προβλήματα και είχε πει ότι ίσως είναι η μόνη περίπτωση ευκαιρία που έχουμε για να θέσουμε ένα ηθικό όριο σε όλα αυτά. Εγώ όταν πήγα στις Ερμές Πολιτείες ε, ε, κατάλαβα ότι ήμουν ο μόνος εκπρόσωπος ε, από, την, από τον ιδιωτικό τομέα και Κατάλαβα ότι ε, στο τέλος ότι κάθε συζήτηση ε, ε, όλοι γυρνούσαν στρέφοντα προς εμένα γιατί έλεγαν «Οκ, πρέπει να μας πει ο Πολ εάν, ποιος θα είναι ο οικονομικός αντίκτυπος». Ε, στην αρχή είχαμε ξεκινήσει βέβαια με τους στόχους της ε, χιλιετίας ε, και είχαμε πει ότι σε 15 χρόνια θα κάναμε μια προσπάθεια για να απαλληφθεί ένα μεγάλο κομμάτι της φτώχειας. Το 2000 προχωρήσαμε στο σχεδιασμό των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και βλέποντας τους ευρύτερους αυτούς στόχους δεν θα εκπλαγεί κανείς βλέποντας ότι ο ιδιωτικό τομέα ε, θεωρείται κεντρικό στοιχείο. Για να λειτουργήσει καλά η κοινωνία θα πρέπει ε, και τα μέλη της ε, να λειτουργήσουν καλά και θα πρέπει και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν καλά γιατί οι επιχειρήσεις θέλουν βιώσιμη ανάπτυξη και έχουν βιώσιμη ανάπτυξη εάν το business model είναι βιώσιμο. Χαίρομαι λοιπόν γιατί ενώ στους στόχους της ε, οι εταιρικέ σχέσεις ε, ήταν μάλλον μία μικρή σκέψη ε, στους 17 καινούριου στόχους βλέπουμε ότι τουλάχιστον οι μισοί δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη συνεργασία και της επιχειρηματικής κοινότητας. και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να οδηγηθούμε σε βιώσιμη ανάπτυξη. Το άλλο θέμα είναι ότι οι στόχοι βιώσιμης ε, ανάπτυξης ε, μπορεί να κοστίσουν 3 με 4-3 ε, δολάρια. ακούγονται πολλά τα χρήματα, αλλά στην ουσία δεν είναι. Η πραγματικότητα μας λέει, όπως έλεγε και ο Τζέφρι προηγουμένως, ότι εάν δεν, δεν είμαστε δραστήριοι όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ε, ο λογαριασμός θα είναι πολύ πιο βαρύς. Μπορεί βέβαια κανείς να στραφεί εναντίον των επιχειρήσεων να πει ότι δεν έκαναν καλά αλλά νομίζω ότι όταν ε, οι οικονομικοί νόμοι στρέφονται εναντίον μας, όλο και περισσότεροι ε, σκέφτονται να ακολουθήσουν έναν άλλο δρόμο. 9% του παγκοσμίου ΑΕΠ ε, κοστίζουν ε, οι πόλεμοι. 3% ε, κοστίζει η έλλειψη ή μείωση βιοπικιλότητας, το κόστος χαμένων ευκαιριών, η έλλειψη ίσων δικαιωμάτων σύμφωνα με το φύλλο, η ελλειπής πρόσβαση ε, των γυναικών ε, στην δουλειά μπορεί να σημαίνει περίπου ένα 15% του συνολικού ε, ΑΕΠ ε, χαμένες ε, μέρες, χαμένες ευκαιρίες μπορεί να σημαίνουν 10 με 12% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια ε, κατάσταση ε, όπου οπωσδήποτε θα πρέπει να απαλείψουμε την φτώχεια με έναν τρόπο συνεκτικό και βιώσιμο και με έναν τρόπο που θα έχει τον λιγότερο δυνατό οικονομικό αντίκτυπο δυστυχώς, ε, ευτυχώς έχουμε ε, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ως οδικό χάρτη. Αυτό που είδαμε όταν συζητούσαμε για θέματα κλιματικής αλλαγής στο Παρίσι, ε, είδαμε ότι γενικώ οι, οι κυβερνήσεις αλλά και ο ιδιωτικός τομέας μέσω των εκπροσώπων που ήταν παρόντες στο Παρίσι συζητούσαν για την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών. Επίσης όλοι ανέφεραν ότι είναι μεγάλο το κόστος και θα είναι μεγάλο το κόστος εάν ε, δεν απανθρακοποιήσουν την λυσίδα παραγωγής τους. Είδαμε λοιπόν στο Παρίσι ότι ε, όλοι, μεταξύ των οποίων και οι εκπρόσωποι των ε, υπεύθυνων εταιριών και επιχειρήσεων. Ε, είδαμε, λέω, όλους να λένε ότι θα πρέπει να βρούμε νέα βιώσιμα μοντέλα ανάπτυξη. Κατανοούμε ότι ε, ίσως οι 17 στόχοι δύσκολα γίνονται κατανοητοί από τις επιχειρήσεις. Ίσως είναι εύκολο να μιλήσει κανείς για την κλιματική αλλαγή γιατί μιλά για ένα συγκεκριμένο θέμα. Ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο να μιλήσει κανείς για 17 ξεχωριστούς ε, στόχους και να μιλήσει για αυτούς τους στόχους και να πείσει για αυτούς τους στόχους επιχειρηματίες οι οποίοι προσπαθούν να παραμείνουν ε, ε, στην δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε την Small Brown ε, να ε, είναι επικεφαλής ε, της Επιτροπής των Εθνών για τα θέματα αυτά. Εκεί έβαλε επιχειρηματίες από μεγάλες και μικρότερες επιχειρήσεις από το UN Global Compact κλπ. Δούλεψαν αυτοί οι άνθρωποι για ένα-ενάμιση χρόνο και παρήγαν μία, και το λέω αμερόληπτα, καλή έκθεση η οποία κάνει μία προσπάθεια να βοηθήσει την ε, ε, κοινότητα των επιχειρήσεων να ενσωματώσουν στα business plan τις, ε, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Γίνεται αναφορά στην ενέργεια, στο, στα διάφορα υλικά, στην γεωργία και στα, στην ενέργεια. Εδώ βλέπουμε τέσσερα hot spots τα οποία ε, τα οποία διαθέτουν, στα οποία συμμετέχουν επιχειρήσεις που διαθέτουν μεγάλη ε, τεχνογνωσία. Τακτοποιήσαμε δε και κάποιους στόχους ενδιάμεσους μέχρι το 2030 και είπαμε ότι περίπου 12-3 ε, ε, δολάρια θα μπορούσε ε, να αντιπροσωπεύσει ή να αντιπροσωπεύσουν οι νέες ευκαιρίες οι οποίες θα ανοίξουν, οι νέες δουλειές, οι θέσεις απασχόλησης οι οποίες θα δημιουργηθούν. Έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να το κάνουμε αυτό και βεβαίως για να το επιτύχουμε θα πρέπει να έχουμε μαζί μας και του, τις επιχειρήσεις. Εγώ ε, ονειρεύομαι ε, μια διαδικασία όπου οι ίδιες ε, οι επιχειρήσεις στρέφονται, θα στρέφονται όλο και περισσότερο προς τους μετόχους και μαζί να βρίσκουν νέα στοιχεία. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο Νομίζω ότι ε, η πρώτη ερώτηση που πρέπει να θέσουμε είναι γιατί αυτές οι επιχειρήσεις ε, ε, κάνουν αυτές τις προσπάθειες. Μα γιατί καταλαβαίνουν ότι, ότι πλέον δεν υπάρχει χρόνος και επίσης όλες οι επιχειρήσεις αυτές μέχρι τώρα έχουν δουλέψει με βράχοι πρόθεσμους στόχους και είναι μια καλή ευκαιρία να ε, ε, σκεφτούν πιο μακροπρόθεσμα. Σε πρώτη λοιπόν φάση ε, εμείς θεωρήσαμε ότι μια ομάδα 1500 διευθυνών των συμβούλων θα ήταν μια καλή αρχή έτσι ώστε να μιλήσουμε για την αρχή της, για την τροποποίηση μάλλον της αλυσίδας αξιών και ε, επίσης ε, υπάρχει και μια μεγάλη ε, παγκόσμια πρωτοβουλία για την σπατάλη ε, την διατροφική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, αν δεν το συνδυάσει κανείς ε, και με την, το οικολογικό ήχρον διατροφικών αυτών ειδών που σπαταλιούνται, τότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη σημασία παίζει όλη αυτή η διαδικασία. Επίσης, άλλες διαδικασίες και πρωτοβουλίες για τη χρήση γης, άλλες πρωτοβουλίες για, τις, για τα δάση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πάρα πολλές ε, πρωτοβουλίες από πλευράς των επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων έτσι ώστε ε, να δημιουργηθεί ένα καλύτερο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Εγώ ε, χτες ήμουν στο Παρίσι γιατί πιστεύω ότι έφτασε η ώρα της Ευρώπης πέρα από κάποιες μικρές λεπτομέρειες, ε, μια μικρή λεπτομέρεια ότι εγώ δηλαδή είμαι Ευρωπαίος, πέρα και από τις ε, προκλήσεις που έχουμε αντιμετωπίσει, πραγματικά εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε να επικρίνουμε την ελληπή λειτουργία του συστήματός μας εάν εμείς δεν κάνουμε ε, μια ε, σημαντική προσπάθεια. Γι' αυτό τώρα είμαι στις Βρυξέλλες, γι' αυτό πριν ήμουν ε, στην Ουάσιγκτον εν ώψη της συνάντησης των G7 για να τους πείσω για κάποια πράγματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Όλα, όλα είναι δυνατά και μπορούμε να επιτύχουμε τη σωστή λέση. Εδώ στις Βρυξέλλες νομίζω ότι έφτασε μια πολύ μεγάλη ώρα. Εγώ ασχολούμαι εδώ και 16 χρόνια με τα θέματα αυτά. Βλέπουμε ε, ότι πλέον μεταξύ της Ευρώπης ε, και της ε, Κίνας υπάρχουν πολύ καλές σχέσεις. Έχουμε την ευρωπαϊκή οικονομία η οποία ανακάμπτει σιγά σιγά και επομένως θα δώσει και λίγο μεγαλύτερο ζωτικό, περισσότερο ζωτικό χώρο από ό,τι τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώ ε, ένα από τα... είχαμε τη Συμφωνία των Παρισίων, δυστυχώ ε, ένα από τους μεγαλύτερου αποφάσισε να φύγει από την συνολική εικόνα. Ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι ε, έχουμε πρόσφατα τις γαλλικέ εκλογές με τις εξελίξεις που γνωρίζουμε όλοι. Είχαμε πρόσφατα και τις ολλανδικές εκλογές στη χώρα μου Ε, και όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έφτασε η ώρα της Ευρώπης ε, και ο Τζέφρι είπε προηγουμένως και συμφωνώ ε, ότι αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης είναι λίγο απογοητευτικό γιατί αναφέρεται μονάχα στα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Τι δεν μπορούμε, τι, τι δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Εάν δει κανείς ε, αν δει κανεί το προσχέδιο για του ε, στόχου βιώσιμη ανάπτυξης είναι τόσο μικρή που ντρέπομαι που είμαι Ευρωπαίο. Έχουμε λοιπόν ε, περιθώρια πολλά για βελτίωση. Έχουμε τώρα ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για την ε, κυκλική οικονομία. Η Έλλην Μακάρθορ ε, έχει ξεκινήσει ένα τέτοιο ε, πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από μόνο του το πρόγραμμα αυτά μπορεί να αυξήσει ένα 1-3 δολάρια το, το ΑΕΠ. Εάν δεν βάλουμε στην, λάβουμε υπόψη μας και τους ωκεανούς, ε, τότε καταλαβαίνετε ε, ε, πόσο περιθώρια έχουμε. Ένα δολάριο το οποίο επενδύεται σε τρόφιμα αποδίδει 17. Ένα δολάριο το οποίο επενδύεται στην, σε υγειονομικά προγράμματα αποδίδει 6 δολάρια. Έφτασε η ώρα να δούμε και πόσο αποδίδουν και τα χρήματα τα οποία επενδύουμε στην ενέργεια. Νομίζω ότι ε, εμείς ε, ε, ξέρουμε αυτά τα πράγματα στην Ευρώπη και νομίζω ότι είμαστε εμείς που είμαστε πιο κοντά στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Έφτασε η ώρα να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να γίνουμε παράδειγμα. Η Ευρώπη μπορεί να δημιουργήσει ένα καλό περιβάλλον και για τους υπόλοιπους, έστω και αν έχουμε προβλήματα σαν αυτά που είδαμε πρόσφατα. Ε, παρά τα προβλήματα, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο, αλλά ε, υπάρχουν δύο-τρία πράγματα τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε. Πιστεύω ότι ε, δεν υπάρχουν επικεφαλής επιχειρήσεων που ε, να μην θέλουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Νομίζω ότι αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης ε, θα πρέπει να σταματήσει. Αλλά πώς είναι δυνατόν εμείς να ε, θέσουμε κάποια όρια στους ανθρώπους αυτούς έτσι ώστε να προχωρήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί βλέπουμε ότι όταν έχουμε ε, μόνο, όταν έχουμε ε, ε, χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίες βλέπουν μόνο το βράχι πρόθεσμο κέρδος, βεβαίως είναι κάτι κακό. Επομένως θα πρέπει τις χρηματαγορές να τις βάλουμε πάλι σε μια μακροπρόθεσμη πορεία. Επίσης ε, είναι αλήθεια ότι κάποιοι είναι καλύτεροι από άλλους, το έχουμε πει, αλλά ε, νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε ένα οικονομικό σύστημα όπου ε, θα είναι καλή και η επιστροφή όσον αφορά το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κεφάλαιο. Ας πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντική, σημαντικό θέμα το να βάλουμε, ε, να βάλουμε μια τιμή ε, στο, ε, στη διοξίδιο του άνθρακα και έτσι να κατανοήσουμε καλύτερα ε, ε, τι, ποιο είναι το διακύβευμα Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, ιδίω ε, όταν η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση βρίσκεται πρώτων πυλών. Ε, έχουμε τη ρομποτική, έχουμε την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει να τα δούμε ε, με βάση και τα διαφορετικά κοινωνικά συμβόλαια του ιδιωτικού τομέα. Νομίζω ότι είναι πολλές ε, οι υπεύθυνε εταιρείε ε, οι οποίες μπορούν να συμπορευτούν με αυτές τις αρχές. Απλώς πρέπει να βρει κανείς στην αρχή μια, έναν αριθμό σημαντικό, μια κρίσιμη μάζα η οποία θα ξεκινήσει την διαδικασία. Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ. Ah, um, uh, thank you, Ευχαριστώ, Πολ. Μας έχει τελειώσει ο χρόνος, αλλά επειδή ζητήσατε το λόγο, σας δίνω ένα λεπτό. Παρακαλώ. 30 δευτερόλεπτα χρειάζομαι ε, και άλλα 30 δευτερόλεπτα για την απάντηση. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ να μας μιλήσετε για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Πολύ σύντομα αναρωτιέμαι, υπάρχει κάποιο ε, παράδειγμα, κάποιο υπόδειγμα στον κόσμο ή στην Ευρώπη. Υπάρχει κάποια χώρα ε, στην οποία μπορούμε να στραφούμε. Η Κολομβία. Η τέλεια απάντηση. Το ίδιο ισχύει με τις επιχειρήσεις. Ε, εργάζονται σε στεγανά. Το ίδιο ισχύει και για τις κυβερνήσεις. Ενώ ε, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ε, είναι σκορπισμένοι στα διάφορα υπουργεία. Εάν λοιπόν έχει κανείς κάποιο πρόγραμμα σε υπουργικό επίπεδο, μάλλον αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει κανείς. Όταν κάποιος ε, φτιάχνει ένα εργοστάσιο στην ε, Κολομβία. Ε, λένε, ωραία, εγώ χρειάζομαι ντομάτες, εσύ χρειάζεσαι ντομάτες, τι να κάνουμε, να συνεργαστούμε, να δούμε τι κάνει το ΦΑΡΚ, να δούμε τι κάνουν τα σούπερ μάρκετ. Ε, γιατί να μην το κάνουμε σε μια περιοχή η οποία κατά τα άλλα ε, θα ήταν αποψηλωμένα δάση. Να φροντίσουμε να έχουμε 50% γυναίκες, να έχουμε ισότητα των δύο φίλων στη διαδικασία αυτή. Επίσης, ε, να εξασφαλίσουμε επαρκές εισόδημα για τους ανθρώπους αυτούς, ώστε να μην έχουμε ε, ε, δουλεία ή εργασία παιδιών. Έτσι λοιπόν εκεί τα σκέφτονται αυτά συνολικά και φροντίζουν την συμμετοχή όλων των παραγόντων και έτσι καταλήγουν σε καλά αποτελέσματα. Και στην εποχή διαφάνειας που ζούμε σήμερα, πολύ λίγα μέρη υπάρχουν όπου να μπορεί να κρυφτεί κανείς. Ε, εγώ τώρα πια απλά πάω και αγοράζω την Financial Times, όπου βλέπω όλα τα στοιχεία για τις εταιρείες. Οι διαφανείς καιροί λοιπόν που ζούμε επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και εάν τα κάνει κανείς αυτά θα πετύχει πολύ καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ, Τζέφρι. 30 δευτερόλεπτα. Δύο γρήγορες παρατηρήσεις. Αν κοιτάξουμε το ευρετήριο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που ε, εκπονεί η ομάδα μου για τα Ηνωμένα Έθνη, θα δείτε στην κορυφή του καταλόγου τους στόχους που ταιριάζουν καλύτερα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη ε, βρίσκει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνική ένταξη. Στην κορυφή του καταλόγου βρίσκονται οι σκανδιναβικές χώρες, ε, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία. Βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου στις περισσότερες ε, κατηγορίες. Η Γερμανία επίσης τα πάει πολύ καλά. και θα έλεγα ότι όλη η Ευρώπη μπορεί να πετύχει όλους τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Όσον αφορά όμως τα εθνικά σχέδια δράσης, πάλι θα έδειχνα την Νορβηγία, τη Σουηδία, όπου υπάρχουν ισχυρές κυβερνητικές δομές. Λένε ότι αυτή είναι εθνική μας στόχη. Η Γερμανία έχει κάνει πολύ καλή δουλειά όσον αφορά την ενσωμάτωση ε, των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης ε, στο πλαίσιο βιωσιμότητας. Οι άλλες χώρες όχι τόσο πολύ. Και τέλος, όσον αφορά τις εξελίξεις αλλού, καθυστερούν. Δεν βλέπουμε προγραμματισμό με στόχο την επιτυχία. Και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο βέβαια έχουν ακόμα δουλειά να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζέφτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας σήμερα. Σας ευχαριστούμε και για την παρουσίαση σας εδώ σήμερα και να δώσουμε το λόγο πάλι στην Πρωθυπουργό τη Νορβηγίας για να κλείσει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήλθατε να μα ακούσατε. Ελπίζω να σας δώσαμε έμπνευση για να εργαστείτε για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Νομίζω ότι ο βουλευτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια πρέπει να τονίσω πόσο σημαντικοί είναι οι βουλευτέ και πώς ε, πραγματικά καλούν τις κυβερνήσεις να λογοδοτήσουν όσα κάνουν. Φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διαφορετικό από τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά ίδιο είναι το καθήκον σας και η δουλειά σας. Ελπίζω λοιπόν να προωθήσετε και να εντάξετε στην δουλειά σας τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ.